Hello everyone, good afternoon. Καλή σας μέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλωσορίζω την προσκεκλημένη μας εδώ για αυτήν την ε, έκτακτη συνεδρίασή μας, την Επίτροπο κ. Πιενκόφσκα. Και πολύ χαιρόμαστε που είναι μαζί μας εδώ σήμερα. Την ευχαριστούμε που ανταποκρίθηκε τόσο γρήγορα στο αίτημά μα για να λάβει χώρα η συνάντηση αυτή, προκειμένου να συζητήσουμε τη συνέχεια που δίνεται στι συστάσεις της ε, ΕΜΙΣ, όσον αφορά τι δικές της αρμοδιότητε, βέβαια. Έχουμε σε 16 γλώσσες διερμηνία και έχετε τα έγγραφα ηλεκτρονικά στη διάθεσή σα, στην ιστοσελίδα μας. Ε, μεταδίδεται και στο διαδίκτυο η συνάντηση αυτή. Κύριε Βιακόφσκα, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Φυσικά, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Είναι πολύ θετικό που μπορούμε να συζητήσουμε... αυτό το μικρόφωνο δουλεύει καλύτερα. Ναι, έλεγα λοιπόν ότι είναι πολύ καλή ευκαιρία που έχουμε προκειμένου να σας ενημερώσω σήμερα για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από πλευράς μας μετά την έγκριση των συστάσεων της Επιτροπής σας έμεις πριν από ένα χρόνο περίπου. Ευχαριστούμε πολύ για τις δικές σας εργασίες, για την προετοιμασία δηλαδή των συστάσεων αυτών. Και για τις συστάσεις αλλά και για την στήριξή σας στο δικό μου έργο. Οι συστάσει σας φυσικά και μα πιέζουν όλους και την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο αλλά και βέβαια πιο σημαντικό τα κράτη-μέλη. Μας πιέζουν όλους να αλλάξουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εργαζόμαστε αλλά επιταχύνουν επίσης και την έγκριση νομοθετικών μέτρων. Τώρα η ευθύνη είναι επιμερισμένη μεταξύ μας προκειμένου να υλοποιήσουμε τις συστάσεις σας. Και εγώ και οι υπηρεσίες μου κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φέρουμε αποτελέσματα. Έχουμε προχωρήσει όσον αφορά τις δοκιμές, τη δέσμη δηλαδή για εκπομπές υπό πραγματικές συνθήκες, για την έγκριση τύπου επίσης, ήδη από το Σεπτέμβριο που μας πέρασε. Επίσης έχουμε προωθήσει και τα νέα μέτρα την παγκόσμια αναρμονισμένη διαδικασία εργαστηριακών δοκιμών. Πρόκειται για αριστηριακέ βέβαια δοκιμέ, αλλά πάντω γίνεται βελτίωση στι μετρήσει όσον αφορά τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα και την κατανάλωση καυσίμων. Επίσης έχουμε ετοιμάσει κατευθυντήριες γραμμές που έχουμε συζητήσει για την έγκριση τύπου από πλευράς των εθνικών αρχών και είμαστε στο τελευταίο στάδιο και όσον αφορά το RDE, δηλαδή τη δέσμη για εκπομπές υπό πραγματικές συνθήκες και όσον αφορά το δεύτερο τμήμα του WLTP που είναι η Παγκόσμια Ενωμένη Διαδικασία Εργαστηριακών Δοκιμών. Ετοιμάζουμε επίσης και την ψηφοφορία στην Τεχνική Επιτροπή την Άνοιξη μετά από διαβούλευση με την κοινή γνώμη. Θέλουμε περισσότερη διαφάνεια στο σύστημα και προτείνουμε οποιοδήποτε εγκεκριμένο εργαστήριο και τεχνική υπηρεσία να μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την επιλογή οχημάτων και την εκπόνηση δοκιμών. Επίσης, οι αρχές για την έγκριση τύπου πρέπει να δημοσιεύουν τα αποτελέσματά τους. Στην τέταρτη πράξη RD αλλάζουμε τη μεθοδολογία όσον αφορά την εκτίμηση των εκπομπών και θα προτείνουμε να είναι υποχρεωτικές για όλα τα νέα οχήματα και τα φορτηγάκια. 26 Ιανουαρίου τώρα. Δημοσιεύσαμε λεπτομερείς πληροφορίες όσον αφορά την κατάσταση πραγμάτων για τα μέτρα ανάκλησης στις διάφορες χώρες μέλη. Το Φεβρουάριο αφιερώσαμε επίσης μάλλον το Φεβρουάριο ε, ε, ζητήσαμε και εγκρίναμε την ε, πλατφόρμα με πληροφορίες όσον αφορά την ανάκληση οχημάτων, η οποία θα ενημερώνεται τακτικά. Έτσι θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε καλύτερα τις έρευνες που γίνονται σε εθνικό επίπεδο και τις δυνατότητες που υπάρχουν για μέτρα παρακολούθησης. Και τέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, έχουμε ξεκινήσει και διάφορες διαδικασίες επί κατά κάποιων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωση, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είτε δεν επέβαλαν ε, τις κατάλληλες κυρώσεις στις αυτοκινητοβιομηχανίες τους, είτε επειδή δεν τηρούν τους κανόνες όσον αφορά τις εκπομπές η Ιταλία για το Fiat 506 για παράδειγμα, Euro 6 diesel, αλλά στείλαμε και επιστολές με κοινοποίηση στη Γερμανία, την Ελλάδα, το Λουξεμβούργο, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αναλύουμε τις τελευταίες πληροφορίες που μας ήρθαν από αυτές τις χώρες μέλη. Η τελευταία χρονιά είχε πολλή δουλειά για μας. Έχουμε προχωρήσει σε πολλά πράγματα, σε άλλα κοντεύουμε να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες. Πάντως το κύριο ε, το κύριο κατόρθωμά μας είναι ότι συμφωνήσαμε για το πλαίσιο. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μας, γιατί θα μας επιτρέψει να ελέγχουμε στην αγορά τα οχήματα όπως θέλουμε και στη συνέχεια να υπάρχει η ανάκληση κυρώσει από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρέπει επίση να υπογραμμίσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τη δικιά του την πλευρά έχει κάνει καταπληκτική δουλειά και σα ευχαριστούμε γι' αυτό. Όπω τόνισε και η Επιτροπή σα, εμεί, οι χώρε μέλη πρέπει να αναλάβουν ευθύνε. Για παράδειγμα, όσον αφορά τον εξοπλισμό retrofitting για τα οχήματα και τα λεωφορεία, τον εξοπλισμό δηλαδή, δεν υπάρχει νομική βάση σήμερα. Θα μπορούσαμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε και θα το κάνω το JRC προκειμένου να γίνονται περισσότερο σε βάθος ε, αναλύσεις τεχνικές για τον εξοπλισμό των οχημάτων και έτσι να μπορούμε να έχουμε καλύτερες πληροφορίες, κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει. Το ίδιο ισχύει και για το περίφημο Monkey Gate. Όπως ξέρετε, η ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι πολύ περιοριστική στον κόσμο όταν πρόκειται για την προστασία των ζώων και τις δοκιμές, τα πειράματα που γίνονται με ζώα. Και οι χώρες μέλη είναι που πρέπει να διασφαλίσουν ότι θα ισχύει αυτό. Από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής πάντως έχουμε ακούσει ε, τι ζητάτε. Την ανεξαρτησία των επιστημονικών σωμάτων και θα κάνουμε σύντομα μία πρόταση σχετικά. Η κυρία Τάισεν δουλεύει από αυτού, η Επίτροπος Τάισεν. Και τώρα κάτι ακόμα που πιστεύω είναι σημαντικό. Ποιο είναι το επόμενο βήμα. Γιατί όλοι πρέπει να κοιτάμε προς το μέλλον. Όλοι συνειδητοποιούμε ότι γίνονται μεγάλες αλλαγές στην αυτοκινητοβιομηχανία. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε και το δεύτερο πακέτο κινητικότητας που θα εγκρεθεί το Μάιο και βάσει αυτού θα ετοιμάσουμε και εμείς ε, μια δικιά μας πρόταση για την συνδεσιμότητα και την αυτόματη οδήγηση. Το πακέτο αυτό θα παρουσιάσει ένα πλαίσιο για αυτά τα ζητήματα και όπως συμβαίνει πάντα με τέτοια θέματα θα ασχοληθούμε και με τις κοινωνικές ε, διαστάσεις. Στηρίζουμε επίσης και την ε, πρόταση να πάμε προς οχήματα μηδενικών εκπομπών. Σε αυτό βέβαια η τεχνολογία θα μας βοηθήσει. Θα πάρει κάποιο χρόνο, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε, να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας και όχι να είμαστε πίσω και απλώς να αντιδράσουμε στις τεχνολογικές αλλαγές που θα λάβουν χώρα κάποια στιγμή. Γιατί η τεχνολογία αυτή μπορεί να συνεισφέρει ε, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην έχει πια εκπομπές άνθρακα. Εμείς ξεκινήσαμε και με την πρωτοβουλία μας ε, για τις μπαταρίες που είναι μια εμβληματική πρωτοβουλία για την παραγωγή μπαταριών. Τον Νοέμβριο επίσης εγκρίναμε ένα πακέτο για καθαρή κινητικότητα για να μειωθούν ακόμα περισσότερο οι εκπομπές ε, ρηπογόνων ουσιών στον αέρα που καταστρέφουν την υγεία. Λοιπόν, δεν έχει τελειώσει το δικό μας έργο. Το έργο της δικιάς σας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής της ΕΜΙΣ μπορεί να τελείωσε, αλλά εμείς συνεχίζουμε και προσβλέπουμε σε παρετέρω συνεργασία μαζί μας τους επόμενους, πώς είναι, 18 περίπου μήνες στηριζόμαστε σε εσά για τις προτάσεις και τις πρωτοβουλίε που έχουμε αναλάβει. Σας ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε ό,τι ερωτήσει έχετε. Ευχαριστούμε κυρία Επίτροπε και τώρα θα ξεκινήσουμε με τον πρώτο γύρο ερωτήσεων. Ξεκινάμε με τους ε, συντονιστές. Ε, πρώτο ο κύριος Γκίζεκε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Μπιενκόφσκα που ήρθε σήμερα στην Επιτροπή μας. Η Επιτροπή ΕΜΙΣ και η Επιτροπή ΕΝΒΗ έχουν ε, μεγάλη χαρά που είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Έχουμε εργαστεί εντατικά μεταξύ μας ε, τους τελευταίους μήνες και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που οι συστάσεις μας ε, θα βρουν εφαρμογή στην πολιτική της Κομισιόν και στην πραγματική νομοθεσία. Στο θέμα της εφαρμογής ε, των συστάσεων της Επιτροπή μας ε, μιλήσατε για το πακέτο, για τον εξοπλισμό, μιλήσατε για την ανάγκη να έχουμε πιο καθαρή ατμόσφαιρα, αλλά και μιλήσατε και για τον γεγονός ότι θέλουμε να εμποδίσουμε παραβάσεις όσον αφορά στα όρια εκπομπών. Επίσης, θέλουμε να έχει ουδετερότητα η τεχνολογία. Θεωρώ ότι αυτή η αρχή είναι ιδιαίτερα σημαντική. Και πραγματικά η τεχνολογία χρειάζεται ουδετερότητα. Η πρόταση του Νοεμβρίου για το διοξίδιο του άνθρακα αφορά στα δημόσια χρήση οχήματα. Υπάρχει ένα σύστημα benchmark συγκρισίμων κριτηρίων δηλαδή, τα οποία θα μας βοηθήσουν να πετύχουμε τις τιμές όρια. Έτσι λοιπόν αναρωτιέμαι αν τελικά είναι ουδέτερη είναι η τεχνολογία. Και αν θέλουμε να μιλάμε για ουδετερότητα της τεχνολογίας, ε, γιατί τελικά η Κομισιόν ασχολείται με μια παλιά τεχνολογία θα πρέπει να υπάρξει ανταγωνισμός μεταξύ των τεχνολογιών. Αυτό είναι ε, ένα από τα σημαντικά συμπεράσματα της εργασίας ε, του Επιτροπής ΕΜΙΣ. Δεν κοιτάμε τις εργαστηριακές τιμέ, αλλά τις πραγματικέ εκπομπές. Σύμφωνα λοιπόν με την πρόταση την νομοθετική, ε, θεωρείται ότι η ηλεκτρική κίνηση είναι σημαντική ε, ενώ δεν αναφέρεται να υπάρχει διαφορά ανάλογα με την πηγή παραγωγής ηλεκτρισμού, όμως πρέπει να δούμε ποιος είναι ο κύκλος ζωής των μπαταριών, από πού προέρχεται το ρεύμα. Έτσι θα μπορέσουμε να δώσουμε και πιο ολοκληρωμένες πληροφορίες στους καταναλωτές ε, για τις πραγματικές εκπομπές. Αυτό το διαπιστώσαμε ε, στο παρελθόν και δεν θέλουμε και στο μέλλον να πάει κάτι στραβά σχετικά. Υπάρχει επίσης ε, το θέμα του εξοπλισμού που είναι ιδιαίτερα αντιφατικό. Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές απόψεις σε κάποιες περιπτώσεις ε, είδαμε ότι είναι δυνατή η μετασκευή, ε, υπάρχουν ε, παλιά ας πούμε οχήματα γύρω πέντε τα οποία μετασκευάστηκαν. Όμως, ποιο είναι το κόστος. Γιατί η βιομηχανία θεωρεί ότι σε μεμονωμένες περιπτώσεις, εντάξει, μπορεί να γίνει, αλλά δεν μπορεί να υπάρχει ε, μαζική παραγωγή. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε αν είναι εφικτό και αν το κόστος είναι ε, αποδεκτό. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντάρλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την Επίτροπο Μπιενκόφσκα που βρίσκεται σήμερα εδώ για να μας ενημερώσει για αυτό το θέμα. Θα ήθελα να ξεκινήσω ε, μιλώντας για τις εκπομπές ε, μονοξιδίου του αζότου. Δυστυχώς ε, έχουμε βιώσει τη συνεχή αποτυχία των ευρωπαϊκών στάνταρ να ελέγξουν αυτές τις τιμές. Έχουμε πρόσφατα τη μελέτη ICCT, είναι οι δοκιμές που έγιναν στο δρόμο και δείχνουν ότι ακόμα και τα, ο στόλος των οχημάτων Euro 6 έχει πολύ υψηλές εκπομπές μονοξιδίου του του αζότου. Ε, πάνω από 400 ε, μιλιγκράμμα ένα χιλιόμετρο αντί για 80. Τι θεωρεί λοιπόν η Κομισιόν ότι πρέπει να γίνει γι' αυτό. Έχει σκοπό να ε, κάνει κάποια αναθερώρηση της σήμανσης ανάλογα με τις δοκιμές των πραγματικών εκπομπών στο δρόμο. Για το ίδιο θέμα επίσης θα ήθελα να ξέρω τι θα γίνει για να δημιουργηθεί ένα αντικειμενικό σύστημα σήμανσης το οποίο θα αντικατοπτρίζει τις πραγματικές εκπομπές, τον πραγματικό κόσμο. Θα ήθελα επίσης να θέσω το θέμα ε, της ε, ανάκλησης οχημάτων. Ε, δυστυχώς ε, φαίνεται ότι η διαδικασία ως τώρα έχει απαράδεκτες ε, καθυστερήσεις. Η Volkswagen έπρεπε να φτιάξει 8,5 εκατομμύρια οχήματα ε, που είχαν συσκευές του 2017, όμως ε, μέχρι σήμερα 2 εκατομμύρια αυτοκίνητα παραμένουν χωρίς επισκευή. Πάνω από δύο χρόνια έχουν περάσει από τότε που μπορέσαμε να ανακαλύψουμε αυτό το σκάνδαλο και συνεχίζουν να υπάρχουν ρηπογόνα οχήματα στους δρόμους παρόλα αυτά. Όσον αφορά τώρα στην απαλλαγή από τις εκπομπές ρηπογόνων ουσιών, η Κομισιόν ελπίζω να φροντίσει να φτιαχτούν αυτά τα οχήματα που δεν συμμορφώνονται, επίσης να τιμωρηθούν τα κράτη-μέλη που δεν έχουν τη θέληση να συνεργαστούν και θα ήθελα να μάθω ακριβώς τι προτίθεστε να κάνετε γι' αυτό. Ευχαριστώ. Η κυρία Βυσινιεύσκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Επίτροπε. Θα συνεχίσω με το σκεπτικό των άλλων σχετικά με το Dieselgate. Στη ΣΥΠΑ, όπως γνωρίζετε, εφαρμόστηκε ένα συγκεκριμένο μέτρο και υπήρξε εξοδικαστική διευθέτηση και η Volkswagen χρειάστηκε να καταβάλει 4,5 δις δολάρια ως αποζημίωση για όλες τις παραβιάσεις. Και αυτό ακριβώς θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εσείς ως εκπρόσωπος θα εισαγάγετε ένα τέτοιο μέτρο κυρώσεων κατά της Volkswagen. την καταβολή ενός χρηματικού ποσού. Γιατί οι πολίτες καταβάλουν το αντίτιμο των παραπτωμάτων της Volkswagen. Ξέρω βεβαίως ότι υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και τα κράτη-μέλη είναι αυτά που επιβάλλουν κυρώσεις. Μπορείτε να λάβετε όμως υπόψη να επιβάλλει χρηματικά ποσά υπομορφή κυρώσεων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της ε, Volkswagen. Ε, μιλήσατε για το Monkey Gate και φυσικά τη στιγμή που γίνονται και έγιναν μάλλον πειράματα με πυθίκους σε θαλάμους ε, αερίων, κοντά στις Βρυξέλλες μάλιστα, αυτό ήταν κάτι που μας εξέπληξε και βεβαίως ήταν κατοικημένη η περιοχή και οι κάτοικοι οι περίοικοι είχαν να υποστούν αρνητικές συνέπειες όπως άσθμα, αναπνευστικά προβλήματα και ούτω καθεξής. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την Επιτροπή ποια μέτρα έχει λάβει για το θέμα αυτό. Τι ακριβώς έχει γίνει και τι μπορείτε να κάνετε εσείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μην συμβεί κάτι τέτοιο και στο μέλλον. Επίσης, θα ήθελα να σας επισύρω την προσοχή στο εξής. Είναι πολύ ανεύθυνο να θέσουμε σε κίνδυνο ορισμένα κράτη-μέλη ως προς τη φήμη τους τη στιγμή που συγκρίνουμε με άλλα κράτη-μέλη όπως το δικό σας. Ξέρετε τι εννοώ. Ως προς την ηλεκτρική κινητικότητα αυτό είναι ένα θέμα που άπτεται της υγείας Επίσης, πώς θα υποστηρίξει η Επιτροπή τα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα τα κράτη-μέλη που έχουν χαμηλό ΑΕΠ, για να εισαχθεί η ηλεκτρική κινητικότητα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Χερμπράντη έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε και ευχαριστώ κυρία Επίτροπε που είσαστε εδώ και σας ευχαριστούμε για τις ε, γραπτές απαντήσεις σας. Έχει μεγάλη σημασία να δούμε πώς προβάλλουμε και υποστηρίζουμε τις νέες τεχνολογίες και δεν είμαστε συντηρητικοί. Θα ήθελα να συγχαρώ την Επιτροπή για όλη την προεργασία για, τις μελλοντικές μας, για τη μελλοντική μας πορεία ως προς τη νέα νομοθεσία. Θα ήθελα να σας συγχαρώ δεν σας καλέσαμε όμως γι' αυτό. Σας καλέσαμε για να μιλήσουμε για τα συμπεράσματα του Dieselgate, ένα από τα μεγαλύτερα βιομηχανικά σκάνδαλα που γνωρίσαμε στην Ευρώπη. Έχω μερικές ερωτήσεις. Πότε θα απαντήσει η Επιτροπή ε, στα ερωτήματα της Επιτροπής περί εκπομπών της ΕΜΙΣ. Πότε θα απαντήσετε στα συμπεράσματά μας. Δεύτερον, το βασικό πρόβλημα είναι τα εκατομμύρια αυτοκινήτων δίζελ που βρίσκονται στους δρόμους και δεν συμμορφώνονται με το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο. Μόνο 7 κράτη-μέλη έχουν υποχρεωτική ανάκληση, 21 κράτη-μέλη δεν έχουν υποχρεωτική ανάκληση. Η Γερμανία ήταν μία από αυτές με τη διάσκεψη περί ντίζελ πέρσι το καλοκαίρι. Όμως το θέμα εστιάστηκε μόνο στη Γερμανία. Όταν η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή επιτρέπει ορισμένα, έναν τύπο μάλλον αυτοκινήτων, τα αυτοκίνητα αυτά μετά πηγαίνουν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άρα γιατί αφήνουμε την γερμανική βιομηχανία να περιορίσει τις ανακλήσεις μόνο για τη Γερμανία. Για μένα αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Κατανοώ τους καταναλωτές. Δηλαδή δεν πάνε στο συνεργείο με το αυτοκίνητο. Γιατί να το κάνουν. Δεν έχουν και κανένα κίνητρο. Πολλές φορές παίρνουν ένα πιο καθαρό αυτοκίνητο, αλλά έχει μεγαλύτερη, μάλλον συγγνώμη, μικρότερη υποδύναμη, γιατί είχε ε, δοκιμαστεί μόνο στην, σε μια περιορισμένη περίοδο, την περίοδο δοκιμών και όχι για να διανύσει εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα. Άρα γιατί οι καταναλωτές να προσφύγουν στα συνεργεία ή στις επιχειρήσεις για αλλαγή οχήματος. Κάτι τέτοιο είχε γίνει στη ΣΥΠΑ. Ξέρω ότι δεν εκπροσωπείται τα κράτη-μέλη, αλλά μας φοβίζει το γεγονός ότι δεν έχει γίνει τίποτα στα κράτη-μέλη. Κανένας δεν έχει, σε κανέναν δεν έχει επιβληθεί χρηματική κύρωση. Μας είπατε ότι δεν έχετε νομική βάση να το κάνετε αυτό, αλλά Πώς συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι στην ατζέντα του Προέδρου Γιούνκερ όταν μιλάς με τους αρχηγούς κρατών και μόνο. Έπειτα, ω προ τις ε, παραβάσεις, πού βρισκόμαστε. Πρέπει να σας διακόψω, λέει η Πρόεδρος, γιατί έχετε υπερβεί τα δύο λεπτά. Μα έχετε φτάσει στα τέσσερα λεπτά και αυτό είναι εις βάρος των άλλων ομιλητών. Όλοι έχουν σοβαρά ερωτήματα. Μπορείτε να επανέλθετε στον επόμενο γύρο ερωτήσεων. Κύριος Eichhout. Εκτός να ε, σας δώσει τα δύο του λεπτά. Έχω και εγώ ερωτήσεις για τις διαδικασίες επί παραβάση. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε που ήρθατε και σας ευχαριστώ και για τις γραπτές σας ερωτήσεις. Για να είμαι ειλικρινής όμως, μερικές φορές έχω την αίσθηση ότι κάποιος άλλος γράφει τις απαντήσεις από ότι όταν έρχεστε εδώ και μας μιλάτε για αυτά. Γιατί είχαμε κάποιες ανταλλαγές απόψεων όπου εσείς ήσασταν σαφέστατοι για το ότι θα υπάρξουν και άλλες διαδικασίες επί παραβάση. Τώρα, όταν διαβάζω τις απαντήσεις, για την ξεκάθαρη ερώτηση κατά πώς θα υπάρξουν και άλλες διαδικασίες ή παραβάση, δεν απαντάτε. Γραπτά δηλαδή δεν μπορείτε να μας πείτε κάτι που μας έχετε πει προφορικά. Και δεύτερον, το πρόβλημα είναι ότι φαίνεται στις απαντήσεις ότι η απαγόρευση των εξοπλισμών που αναστέλουν τους ελέγχους είναι εθνική αρμοδιότητα. Μα Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει προκειμένου να φροντίζει να συμμορφώνονται οι, μέλη, χώρες μέλη με τον Ευρωπαϊκό νόμο. Και ο Ευρωπαϊκός νόμος λέει ότι απαγορεύονται αυτοί οι εξοπλισμοί αναστολής ελέγχων. Οπότε, όταν μια χώρα δεν σέβεται τον Ευρωπαϊκό νόμο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προβεί σε μια διαδικασία επί παραβάση. Κάτι το οποίο δεν κάνετε οι κατευθυντήριες γραμμές σας για τους εξοπλισμούς αυτούς λένε ότι τελικά υπάρχουν πολύ περισσότεροι τέτοιοι εξοπλισμοί που κυκλοφορούν στις χώρες μέλη. Γιατί λοιπόν δεν κάνετε κι άλλες διαδικασίες επί παραβάση κατά των χωρών που επιτρέπουν να χρησιμοποιούνται τέτοιοι εξοπλισμοί. Οι απαντήσεις σας γραπτά πραγματικά είναι πολύ ασαφείς. Η διαδικασία επί παραβάση είναι μια διαδικασία, αλλά έχουμε μηχανήματα τα οποία ρηπαίνουν την ατμόσφαιρα και έχουν τέτοιου εξοπλισμούς. Τι θα γίνει για αυτά. Και τι είναι αυτή η πλατφόρμα ενημέρωση για την ανάκληση οχημάτων. Ποιο είναι ο στόχος μιας τέτοιας πλατφόρμας. Ότι πάλι ωραία και καλά και ευγενικά θα ζητήσετε από τι χώρε μέλη να κάνουν κάτι, χωρίς όμως να επιβάλλετε. Όχι, θα έπρεπε να γίνεται υποχρεωτική αυτή η ανάκληση. Αλλιώς και πάλι κοροδευόμαστε. Δεν νομίζω ότι πρέπει να συνεχίζεται αυτό. Ωραία, δύο λεπτά κράτησε. Τήρησα το χρόνο μου. Ωραία, πολύ θετικό το παράδειγμά σας, λέει η Πρόεδρος κυρία Ικάουτ. Η κυρία Εύη τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Μπιενφκόσκα, σας ευχαριστώ και καλημέρα σας. Και εγώ θα σας υποβάλω ερωτήσεις και ξεκινώ από την πιο σημαντική για μένα. Αφορά τις διαδικασίες επί παραβάση. Καταλαβαίνω βέβαια ότι δεν μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες, αλλά στην περίπτωση αυτή της διαδικασίας επί παραβάση κατά των χωρών που δεν έχουν προβεί σε κυρώσεις αλλά και κατά της Ιταλίας γιατί υπάρχει το μοντέλο Fiat 500 X, το οποίο χρησιμοποιεί παράνομο λογισμικό, από ό,τι λέγεται. Μετά από τόσους μήνες που ξεκίνησε η διαδικασία επί και παρά τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να ορίσουμε αυτό το πλαίσιο των διατάξεων αναστολής, δεν υπάρχει σαφήνεια έτσι ώστε χωρίς αμφισημίες να ε, δούμε κατά πόσο υπάρχει παράνομο λογισμικό για αυτό το μοντέλο της Fiat. Στη συνέχεια ε, υπήρξαν πρωτοβουλίες και σε τοπικό επίπεδο από πολλούς δήμαρχους που απαγορεύουν τα αυτοκίνητα diesel στην πόλη τους, Παρίσι, Μαδρίτη, Ρώμη, Αθήνα και ούτω καθεξής. Μιλάμε λοιπόν για συνοδευτικά μέτρα έτσι ώστε να προστατεύσουμε την υγεία και τον αέρα που αναπνέουμε. Μπορείτε να μας πείτε κατά πόσο θα προωθήσετε πιο συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές που θα βοηθήσουν τους δημάρχους που έχουν αναλάβει αυτές τις πρωτοβουλίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία Μελά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Ε, ευχαριστούμε για την ε, ενημέρωση αυτή. Είχαμε ένα σκάνδαλο το οποίο και κατέδειξε τους κινδύνους από ορισμένους κινητήρες που βλάπτουν λόγω και του εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και των οξυδίων ε, του αζότου, αλλά από την άλλη μεριά έτσι καταστρέφεται και η οικονομία μας σε έναν βαθμό. Οπότε, από τη μια μεριά πρέπει να δούμε την κατασκευή και από την άλλη μεριά τον κινητήρα και την κατασκευή του οχήματος αλλά και τον κινητήρα. Το θέμα είναι πώς δημιουργείται ο ηλεκτρισμός και πώς τον αποθηκεύουμε. Τα ντίζελ θα πρέπει να περιοριστούν όσο γίνεται πιο γρήγορα, όλοι συμφωνούμε γι' αυτό. Η συζήτηση όμως δεν προχωράει αρκετά. Τα οχήματα diesel που κυκλοφορούν παραμένουν, είναι πολλά. Πώς θα τα περιορίσουμε. Κυρία Επίτροπε, έχω την εξής ερώτηση. Τι περιθώρια ελιγμών θα αφήσει στις χώρες μέλη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διαχειριστούν ένα ζήτημα δημόσιας υγείας και βιομηχανικής πολιτικής, εθνικής, όσον αφορά την καινοτομία στους κινητήρες. Ευχαριστώ. Ωραία. Εσείς τώρα να απαντήσετε κυρία Επίτροπε. Ωραία. Θα προσπαθήσω να δώσω τις ε, απαντήσεις που χρειάζεται. Of course, ε, ε, It's okay. It works. Yes. Για την ε, ουδετερότητα της τεχνολογίας ε, φυσικά συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός ε, μεταξύ των διαφορών τεχνολογιών φυσικά. Και γι' αυτό στα διάφορα πακέτα μας και στο πακέτο για την κινητικότητα του Μαΐου, είναι το τρίτο πακέτο, μιλάμε όσον αφορά στα αυτοκίνητα μηδενικών εκπομπών, μιλάμε και για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα αλλά και για τις κυψέλες καυσίμων. Έτσι λοιπόν η οδετερότητα της τεχνολογίας διασφαλίζεται με αυτόν τον τρόπο. Και φυσικά είναι και το θέμα των ε, ηλεκτρικών στυλών, των μπαταριών. Ε, μέσα από το ETS ε, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει ουδετερότητα σε επίπεδο εκπομπής οξυδίων του άνθρακα και άλλων ρηπογόνων ουσιών. Για το γύρο 6 και την κατάσταση σχετικά με αυτό. Ε, γνωρίζουμε το πρόβλημα, αλλά θα πρέπει να επαναλάβω ότι αυτά τα αυτοκίνητα έχουν έγκριση τύπου σύμφωνα με τους παλιούς κανόνες. Με τους νέους κανόνες όλα αυτά θα αλλάξουν για τις ανακλήσεις. Τεράστιο πρόβλημα. Συμφωνώ με πολλούς από εσάς που έχουν ήδη ε, ρωτήσει σχετικά και έχουν μιλήσει για αυτό το θέμα. Και εγώ δεν είμαι ευχαριστημένη φυσικά με το επίπεδο των ανακλήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως μπορεί να γνωρίζετε, έστειλα επιστολή πέρυσι το καλοκαίρι. Και μετά από αυτή, τα κράτη-μέλη που έκαναν υποχρεωτικές ανακλήσεις από τέσσερα έγιναν 7. Πάλι δεν είναι ικανοποιητικό το νούμερο, αλλά τουλάχιστον υπήρξε αντίδραση στην επιστολή μου. Υπάρχουν βέβαια διάφορα επίπεδα, ε, από 92% στη Γερμανία, όπως αναφέρατε, ε, έχουμε μόνο 30% στην Ρουμανία. Υπάρχει διακύμανση δηλαδή. Ρουμανία, Σλοβακία είναι σε χαμηλά επίπεδα. Και αυτό φυσικά δεν είναι αποδεκτό και γι' αυτό θα συνεχίσω. Γιατί η πλατφόρμα, γιατί θεωρήσαμε, θεώρησα ότι με την δημοσίευση των δεδομένων και με την υποχρεωτική υποβολή δεδομένων που πρέπει τα κράτη, που πρέπει τα κράτη μέλη ε, να έχουν, θα υπάρξει μια πολιτική πίεση στα κράτη μέλη. Γιατί σύμφωνα με το νέο σύστημα εγκρίσεων τύπου θα μπορούμε να έχουμε και ευρωπαϊκές ανακλήσεις. Διαφορετική κατάσταση από την, σε σχέση με την τρέχουσα. Όλα αυτά θα μας κάνουν να ασκήσουμε όλο και μεγαλύτερη πίεση στα κράτη-μέλη για να ασκήσουν με τη σειρά τους πίεση στις εταιρείε. Γιατί θεωρώ ότι μια υπεύθυνη εταιρεία, ελπίζω τουλάχιστον, αυτό είναι μια ιδεατή κατάσταση ίσως, αλλά τέλος πάντων μια υπεύθυνη εταιρεία στην πράξη θα προσπαθήσει να βρει υποστήριξη από την πλευρά των εθνικών αρχών. Για παράδειγμα, να ζητήσει την εισαγωγή υποχρεωτικών ανακλήσεων. Προς το παρόν έχετε δίκιο. Η Volkswagen ούτε έκανε ε, κάποια ανάκληση από μόνη της, ε, ούτε συμμορφώθηκε με τα χρονοδιαγράμματα για τις διαδικασίες επί παραβάση. Έχω ξεκινήσει τέτοια διαδικασία για την Ιταλία. Ε, μπορώ να σας στείλω κάποιες λεπτομέρειες επιπλέον, αλλά ούτω ή άλλω έχουμε στείλει μια συμπληρωματική επιστολή για το θέμα αυτό σε 7 κράτη-μέλη. Και βέβαια περιμένουμε, γιατί αυτή τη στιγμή κάνουμε ανάλυση των απαντήσεων των κρατών μελών. Δεν βλέπω κάποια δυσαναλογία ή τέλος πάντων κάποια συμφωνία μεταξύ αυτών που λέω εδώ και όσων υπάρχουν στο χαρτί. Όπως και να έχει, από καμία διαφορά. Δεν ε, καταλαβαίνω ε, γιατί το λέτε. Ούτως ή άλλως ε, είναι μια πιο αναλυτική απάντηση αυτή που δίνω εδώ. Ίσως αν κάνω και μια περαιτέρω ανάλυση, δεν μπορώ να σας πω τώρα, αλλά τέλος πάντων μπορώ να κάνω κάποια συμπληρωματική ενημέρωση όπως αυτή που έχω για την Ιταλία. Τώρα, η αποζημίωση των καταναλωτών. Μάλλον όχι αποζημίωση, τα χρηματικά πρόστιμα. Τώρα θα μιλήσω πολωνικά, γιατί το θέμα αυτό, η ερώτηση έγινε στα πολωνικά. Μάλλον μιλάω αγγλικά. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Γυρίζω στα πολωνικά. Λοιπόν, η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν προβλέπει αποζημίωση για τους ιδιοκτήτες οχημάτων, δηλαδή για τους καταναλωτές, όπως γίνεται στις Ηνωμένε Πολιτείες. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια χρηματικά πρόστιμα, τα οποία έχουν επιβληθεί στους ε, κατασκευαστές αυτοκινήτων. Αυτά μπορούν να τα επιβάλλουν τα κράτη-μέλη. Οι παραβάσεις οι διαδικασίες επί παραβάση τέλος πάντων έχουν ξεκινήσει για χώρες στις οποίες οι εταιρείε δεν έχουν την κατάλληλη διαδικασία και όπου τα χρηματικά πρόστιμα είτε δεν επιβάλλονται καθόλου, είτε δεν επιβάλλονται σωστά, είτε τέλο πάντων δεν υπάρχουν στην εθνική νομοθεσία. Δεν υπάρχει νομοθετικό εργαλείο δηλαδή να ε, υπάρχει συγκεκριμένα για τους ε, παραγωγούς αυτοκινήτων σε αυτές τις χώρες. Άρα, ναι, τα κράτη-μέλη έχουν την ευθύνη για να επιβάλλουν τα χρηματικά πρόστιμα, όμως αυτό που κάναμε εμείς με τις εγκρίσεις τύπου ήταν να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε να μπορούν να επιβάλλουν πρόστιμα μέχρι και 30.000 ευρώ ανά όχημα. Αυτά τα πράγματα μπορέσαμε να τα θεσπίσουμε τον Δεκέμβρη. Τώρα, οι δοκιμές στα ζώα, που τελικά είναι δοκιμές σε ανθρώπων, σε ανθρώπους, αναφέρατε έναν οργανισμό ο οποίος όμως δεν είναι ευρωπαϊκός. Ε, μπορεί να ονομάζεται ευρωπαϊκός οργανισμός κάτι, αλλά δεν είναι ευρωπαϊκός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι επειδή είναι στην Ευρώπη. Αυτή η υπόθεση πραγματικά είναι φρικιαστική για μένα γιατί σχετίζεται και με την αυτοκινητοβιομηχανία αλλά και με δοκιμές, δοκιμασίες σε ζώα που καταλήγουν τελικά να είναι δοκιμασίες σε ανθρώπους. Και υπήρξε μια ανταλλαγή επιστολών με τη γερμανική κυβέρνηση και κατά πρόσωπο ανταλλαγή απόψεων για να μπορέσουμε να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη γιατί αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Τώρα, για την ηλεκτροκίνηση, για τις μπαταρίες, ε, τις κυψέλες καυσίμων κτλ. Είναι ένα θέμα με το οποίο έχω ασχοληθεί πάρα πολύ. Και τώρα, σύμφωνα με τα project του Ορίζοντα 2020, ε, έχουμε υποστήριξη για αυτά τα ζητήματα. Θα είναι σίγουρα όμως και μία από τις προτεραιότητες για τον επερχόμενο προϋπολογισμό. θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ε, μια task force, ε, ένα σχέδιο τέλος πάντων για να μπορέσουμε να προωθήσουμε την ηλεκτροκίνηση και να φροντίσουμε ώστε να γίνεται καλύτερη χρήση των μπαταριών κτλ. Να διευρυνθεί η χρήση τους. Αυτά τώρα βέβαια θα συζητηθούν όταν μιλήσουμε και για τον προϋπολογισμό. Γενικά είναι καλό να έχουμε πόρους για τις υποδομές όχι μόνο για την παραγωγή των ε, προϊόντων, δηλαδή των κυψελών καυσίμων κτλ. Γιατί δεν είναι μόνο η κατασκευή των οχημάτων, είναι να υπάρχει και η κατάλληλη υποδομή για την κατασκευή τους και για τις μπαταρίες ε, στα οχήματα. Τώρα για τα συμπεράσματα της Επιτροπής έμις ε, να έχω ακόμα μία απάντηση να δώσω. Κοιτάξτε, δεν μπορώ τώρα να σας δώσω τη συγκεκριμένη ημερομηνία για το πότε θα απαντήσουμε σε αυτά τα συμπεράσματα της Επιτροπής εμείς. Ε, ως τώρα ασχολούμαστε με τις συστάσεις. Τέλος πάντων, είμαστε έτοιμοι να τα κάνουμε ένα πακέτο και να απαντήσουμε σε μία-μία τις ε, συστάσεις, ε, τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα για τις εκπομπές, ε, για το, ε, για το RDE, τις εκπομπές κατά την πραγματική χρήση των οχημάτων και για όλα αυτά τα ζητήματα. Η δική μου θητεία θα οδηγήσει θα καταλήξει και σε ένα δεύτερο γύρο ανταλλαγών απόψεων μέσα στους επόμενους 18 μήνες δηλαδή. Βέβαια δεν έχω απαντήσει τώρα σε όλες τις ερωτήσεις σας, αλλά θα έχετε και γραπτά κάποιες απαντήσεις. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, το πιο σημαντικό για μένα είναι το θέμα των χαμηλών ποσοστών ανακλήσεων. Νομίζω ότι σίγουρα χρειάζεται να αυξήσουμε την πίεση, γιατί καταλαβαίνετε ε, ατύπως το έχουμε κάνει, αλλά πριν και τις επόμενες εγκρίσεις τύπου θα πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός ανακλήσεων σε κάποια κράτη-μέλη τουλάχιστον. Γιατί αυτά είναι τα κράτη-μέλη στα οποία ο αριθμός των οχημάτων με τις λανθασμένες συσκευές με τις διατάξεις αυτές ε, που αναστέλουν, παρακάμπτουν τους ελέγχους, ε, έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα. Επίσης είχα συνεργασία και με τον Γερμανό Υπουργό. Τώρα που θα έχουμε και την καινούργια κυβέρνηση θα είναι πιο εύκολο, πιο απλό. Όχι, δεν το πιστεύετε. Εντάξει. Όταν υπάρχει μια μόνιμη κυβέρνηση είναι πιο εύκολο να συζητάς μαζί της, έτσι δεν είναι. Δεν είναι τόσο εύκολο. Αυτά ως τώρα. Α, α όχι. Α, κάτι άλλο ακόμα. Όσον αφορά τις αποζημιώσεις και τους καταναλωτές, κάποια άλλη ερώτηση. Το σκάνδαλο αυτό έδειξε και τα όρια των εθνικών διαδικασιών προκειμένου να προστατεύσουν τους καταναλωτές. Γι' αυτό λοιπόν και τώρα εργαζόμαστε, χωρίς να είναι βέβαια μόνο δικιά μου αρμοδιότητα, αλλά με την Επίτροπο Γιούροβα ε, συνεργάζομαι. Και σίγουρα θα προτείνουμε κάτι για συλλογική αποζημίωση των καταναλωτών. Να προβλέπετε δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αυτό το νέο εργαλείο, το νέο μέσο, ώστε έτσι να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο αυτοκινητοβιομηχανίες. Ωραία, νέος γύρος ερωτήσεων, ο κύριος Βίμπ πρώτα. Παρακαλώ. Δύο λεπτά. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Επίτροπε. Έχω την εξής ερώτηση. Το Dieselgate θα κρατήσει πολύ ακόμα. Γιατί εμεί θέλουμε να λυθεί και να λυθεί και σωστά. Όμως αυτό το ζήτημα επιτρέπει να διονύζονται αμφιβολίες για αυτού του είδους τα οχήματα. Και αυτό είναι που ανησυχεί τους καταναλωτές. Η έλλειψη εμπιστοσύνη. Εσείς ε, λοιπόν Πώς βλέπετε το θέμα αυτό του, της μετασκευής των ε, οχημάτων του δημόσιου τομέα, για παράδειγμα. Τι θα κάνετε γι' αυτό. Έχουμε το σχέδιο κανονισμού τώρα για τα καθαρά οχήματα. Πώς θα προχωρήσει. Και αυτό βέβαια συνδέεται άμεσα και με τους εναλλακτικούς τύπους οχημάτων, όπως είπατε. Βεβαίως, θέλουμε καθαρά οχήματα και μπορούμε να δημιουργήσουμε αντίστοιχη νομοθεσία για καθαρά οχήματα, αλλά δεν μπορούμε να νομοθετήσουμε ότι θα υπάρξουν και όλα. Αν χρησιμοποιούν καθαρή τεχνολογία θα έχουν την ίδια ισχύ. Αυτό βέβαια μπορεί να είναι δευτερεύον. Αλλά η ερώτησή μου είναι βασικά κατά πόσο η Ευρώπη μπορεί να στηρίξει τέτοια τεχνολογία. Οι τοπικές αρχές έπειτα. Αυτές είναι που θα φροντίσουν να χρησιμοποιηθεί αυτή η τεχνολογία στα ΙΟΤΑΧΗ. αλλά θα υπάρξουν ε, μηχανισμοί στήριξης οχημάτων που χρησιμοποιούν ε, τέτοιε καθαρές τεχνολογίες. Η κυρία Σάλντεμόζε τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ και εγώ για την τόσο καλή συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα για την έγκριση τύπου, που είμαι σίγουρη ότι θα λύσει πολλά προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, και άλλα χρειάζεται να γίνουν. Είπατε και εσείς δύο ότι πρέπει να πιέσουμε περισσότερο τις χώρες μέλη. Εσείς Είχατε επαφή με τους υπουργούς, με τις πρωτεύουσες απευθείας, εσύ ίδια. Και θέλω επίσης να ξέρω, κάποια αυτοκινητοβιομηχανία ήρθε σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να προσπαθήσει να καταλάβει την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ήρθαν σε επαφή μαζί σας. Θα ήταν καλό κάτι τέτοιο. Ή εξακολουθούν να δείχνουν απροθυμία να συμμορφωθούν με την νομοθεσία. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Φέντελη. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ, κυρία Πίτροπε, που ήρθατε να συζητήσετε μαζί μας αυτά τα σημαντικά πράγματα. Πρώτον, κάτι που σχετίζεται και με άλλες ερωτήσεις, οποίες απαντήσατε γραπτά, ρωτήθηκαν και εδώ, διαδικασίες επί παραβάση. Λέτε στη γραπτή σας απάντηση ότι σκέφτεται ποιο θα είναι το επόμενο βήμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωραία, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για αυτό το επόμενο βήμα και τι θα γίνει με τις διαδικασίες επί παραβάση, τι συνέχεια θα δοθεί. Δεύτερον, βλέπετε ότι όλο και περισσότερες πόλεις απαγορεύουν ή περιορίζουν τέλο πάντων τα οχήματα diesel. Και αυτό είναι καλό για τη δημόσια υγεία, τα περιβαλλοντικά. Αν κάνουμε καλά τη δουλειά μας και βάλουμε τις σωστές προδιαγραφές και τηρούνται οι κανόνες που έχουμε εφαρμόσει, δεν θα χρειαζόταν βέβαια η μία μετά την άλλη πόλη να εμποδίζουν τα οχήματα ντίζελ να κυκλοφορούν σε αυτές για να προστατεύσουν ε, την υγεία των πολιτών τους. Ευχαριστούμε. Δύο λεπτά κύριος τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Έχουμε 35 εκατομμύρια όχι εγώ. Όχι, κύριε Σντάν, είπατε έχει το λόγο, όχι εσείς κύριε Τούρμες. Αν νόμιζα ότι μετά τους φιλελεύθερου παίρνουν το λόγο οι πράσινοι, αλλά φαίνεται όχι. Ε, όχι. Μετά τον κύριο Ντάν είσαστε εσείς. Δύο λεπτά κύριε Ντάν. Τρία λεπτά νόμιζα ότι είχα. Όχι. Έτσι μου είπανε. Τέλο πάντων. Ωραία. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Καλό είναι που σας έχουμε εδώ πάλι. Για τις ε, διαδικασίες δοκιμών. Η Επιτροπή πρότεινε τον Μάρτιο κάποια πράγματα, αλλά έχει υπάρξει καθυστέρηση όσον αφορά την ψηφοφορία κτλ. Τι θα γίνει τελικά για τη διαδικασία της CMV, e την Τεχνική Επιτροπή δηλαδή για τα μηχανοκίνητα οχήματα. Είπατε ότι από 20-10% έχουν μειωθεί κάποιες μετρήσεις. Οι προσδοκίες σας σχετικά με αυτά προχωρούν. Ο παράγοντας δηλαδή συμμόρφωσης από 1,2 σε 1,4 πιστεύετε ότι ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας. και σχετικά με τις συστάσεις της Επιτροπής μας. Φυσικά και θέλουμε προδιαγραφές που να μειώνουν όσο γίνεται περισσότερο τις εκπομπές. Η Κίνα που είναι κάτω από το Euro 6, την προδιαγραφή Euro 6 δηλαδή, παρόλα αυτά οι, τα κινέζικα οχήματα θα μπορούν να πολλούνται στην ευρωπαϊκή αγορά, ενώ τα ευρωπαϊκά οχήματα που δεν θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές για το οξύδιο του αζότου δεν θα μπορούν να πολλούνται στην Κίνα. Και για την ουδετερότητα της τεχνολογίας παραδέχεται η Επιτροπή ότι δεν τα καταφέρει να ανταποκριθεί στον ανταγωνισμό κυρίως με την Κίνα που έχει σαν στόχο τις μηδανικές εκπομπές. Τι θα γίνει και είναι ικανοποιημένη η Επιτροπή για τη νέα πρόταση για τις εκπομπές του του άνθρακα που δεν περιλαμβάνει εντολή για οχήματα με μηδενικές εκπομπές. Ε, σχεδόν δύο λεπτά. Τώρα είναι ο κύριος Τούρμας. Δυόμιση χρόνια είμαστε μετά από το Dieselgate και έχουμε 35 εκατομμύρια νέα οχήματα diesel τα οποία ρηπαίνουν πάρα πολύ. Και η, τα λογισμικά για την αλλαγή των οχημάτων δεν έχει προχωρήσει αρκετά. Οπότε, συμφωνείτε ότι η ενημέρωση των λογισμικών δεν φτάνει για να λυθεί αυτό το θέμα στην μετασκευή. Έπειτα, οι Γερμανοί αποφάσισαν να απαγορεύσουν το ντίζελ. Πολύ καλό για τους Γερμανούς πολίτες, αλλά πολύ κακό φοβάμαι για τους πολίτες στην Ανατολική Ευρώπη αν δεν τους προστατεύσουμε. Γιατί τι θα γίνει, οι Γερμανοί πολίτες τώρα θα πουλήσουν τα οχήματά τους ντίζελ μεταχειρισμένα και ποιος θα τα πάρει, η Ανατολική Ευρώπη. Και θα ρηπανθεί η Ανατολική Ευρώπη για δεκαετίες. Αυτό είναι πολύ εύκολο, αλλά θα έπρεπε να είναι υποχρεωτική η μετασκευή για όλα τα Euro 5 και Euro 6 και η Ένωση Οχημάτων θα έπρεπε να φροντίσει να επιβληθεί αυτή η μετασκευή. Σε κάθε περίπτωση οχημάτων στο οποίο είχε μπει αυτός ο εξοπλισμός αναστολής ελέγχων. Θα ήθελα δηλαδή να μας πείτε ότι επιτέλους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έρθει και θα μας πει ποιοι κινητήρες Euro 5 και Euro 6 μπορούν να μετασκευαστούν. Αλλιώς, σας λέω, είναι σκάνδαλο αυτή η πολιτική της γερμανικής κυβέρνησης. Δεν νομίζω ότι οι πολίτες των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης θα έχουν χρήματα για να αγοράσουν γερμανικά αυτοκίνητα. Εγώ θα μιλήσω από το, μίλησα από το χρόνο του ΕΛΚ. Η κυρία Κάντεμπαχ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ καταρχάς και δεύτερο που είστε σε θέση και έτοιμοι να μας δώσετε αναλυτικές απαντήσεις. Η δική μου ερώτηση είναι λίγο πιο γενική. Σήμερα και μετά από τα όσα είπε και ο κύριος Τούρμες, τονίσατε πολλές φορές ότι πρώτον στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της ιστορινής νομοθεσίας δεν υπάρχει αποζημίωση για τους καταναλωτές, αντίθετα με τις Ηνωμένε Πολιτείες, αλλά αυτό που δεν είπατε ή δεν είπατε επαρκώς είναι ότι δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με παραβίαση των δικαιωμάτων των αγοραστών και των καταναλωτών, αλλά και με παραβίαση του γενικότερου συμφέροντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για το δικαίωμα σε ένα υγιές περιβάλλον και στην σωματική ακαιρεότητα. Ε, υπάρχει μια μελέτη του ΩΣΑ που σύμφωνα με την οποία το κόστος ε, του να μην ασχοληθεί κανείς με το θέμα είναι πολύ μεγάλο. Μιλήσαμε για το κόστος των ανακλήσεων και των μετασκευών, όμως ε, έχετε δει στην Κομισιόν ε, τι γίνεται ε, και σε τι τάξη μεγέθους ανέρχεται το κόστος της μη αντιμετώπισης του προβλήματος. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Γιατί έτσι, αν το γνωρίζατε αυτό, θα ήταν πιο συγκεντρωμένη η προστασία του περιβάλλοντος θα γνωρίζατε πολύ καλά και θα ήσασταν ενημερωμένοι για να προστατέψετε το περιβάλλον και να έχουμε μια πιο και μια καλύτερη ε, υγεία για τους καταναλωτές. Συνεπώς, έχει δει η Ευρωπαϊκή Ένωση πόσα χρήματα ε, θα χαθούν στο μέλλον και από επενδύσεις επειδή έτσι αμελώς έχει ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Ε, τώρα θα μπορέσω να επιτρέψω άλλες τρεις ερωτήσεις, αν υπάρχουν. Ο κύριος Χερμπράντι και η κυρία Εύη θέλουν το λόγο. Ο κύριος Χερμπράντι πρώτα. Πρόεδρε, ευχαριστώ για αυτό το επιπρόσθετο λεπτό. Για τη διαδικασία επί παραβάση. Δεν ξέρουμε ακριβώς πού βρισκόμαστε. Φτάσατε στο επόμενο βήμα ή μελετάτε τις πληροφορίες των κρατών μελών, γιατί αυτό το κάνετε από πέρσι τον Ιούνιο. Άρα η ερώτησή μου είναι γιατί είναι τόσο χρονοβόρα η διαδικασία. Είναι νομικά και τεχνικά περίπλοκη ή από πολιτικής πλευράς ε, υπάρχουν δυσχέρειες ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, ως προς τις βινιέτες που κυκλοφορούν στις πόλεις της Ευρώπης, αν πηγαίνετε ε, διακοπές πρέπει να αγοράσετε βινιέτα από κάθε πόλη ή χώρα. Θα προσπαθήσετε να έχουμε ώστε να έχουμε μία ευρωβινιέτα η οποία να είναι ενιαία για όλους για τις πόλεις που δεν επιτρέπουν τη χρήση δίζελ. Η κυρία Εύη, ευχαριστώ. Θα ήθελα να υποβάλω μία ερώτηση σε σχέση με την τεχνολογική ουδετερότητα. Θα ήθελα να μας πείτε κατά πόσο νομίζετε ότι αυτή η αρχή έμπρακτα είναι κάτι που έχει ξεπεραστεί. Γιατί αν συνεχίσουμε να τασόμαστε υπέρ της ε, τεχνολογικής ε, ουδετερότητας, όπως θέλουν οι συντηρητικοί οι χριστιανοδημοκράτες, τότε δεν θα φτάσουμε πουθενά. Εσείς το είχατε πει και δημοσίως αυτό, ότι τα διζελοκίνητα αυτοκίνητα πρέπει να ξεπεραστούν. Άρα Πέρα από τις ε, δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, εσείς θεωρείτε ότι δεν θα πρέπει να υποστηρίζουμε μία συγκεκριμένη τεχνολογία η οποία μολύνει και θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι πέρα από το πακέτο της κινητικότητας το οποίο δεν είναι φιλόδοξο και άρα να μπούμε σε καθαρές τεχνολογίες. Ευχαριστούμε. Λίγη και αυτός ο γύρος των ερωτήσεων. Μπορείτε να απαντήσετε, κυρία Επίτροπε. Θα αρχίσω με τις παραβάσεις. Κατανοώ αυτό που λέτε. Μελετούμε τις απαντήσεις, γιατί είναι ένα τεχνικά δύσκολο ζήτημα και Προσπαθούμε να συνεργαστούμε με τον Επίτροπο Βέλα, ο οποίος ασχολείται με τις διαδικασίες επί παραβάση και για τη μόλυνση του αέρα. Δεν θα μπορέσω να σας δώσω χρονοδιάγραμμα, σαφές χρονοδιάγραμμα για τους επόμενους μήνες. Σε πάση περιπτώσει θα σας πω πότε θα φτάσουμε στο επόμενο βήμα για τις ε, παραβάσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα είναι λεπτομερές, αν θα σας ικανοποιήσει, αλλά θα σας στείλουμε ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα. Μην, ε, μην με συγχαίρεστε γιατί δεν ξέρω, μην με χειροκροτάτε γιατί δεν ξέρω τι θα σας δώσω ακόμα. Ο, ο βοηθός μου, ο Κάρστεν, δεν επιτρέπει τίποτα όπως τον ακούτε. Εν πάση περιπτώσει θα σας πω ποια θα είναι τα επόμενα βήματα γιατί είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, πρόκειται για τεχνικά δύσκολα ζητήματα και δεύτερον προσπαθούμε να συμβαδίσουμε με τον Επίτροπο Βέλα και τις δικές του υπηρεσίες γιατί ασχολείται με τις παραμβάσεις ως προς τη μόλυνση του αέρα. Θα μιλήσω πάλι στα πολωνικά. Υπάρχουν δύο μέσα τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε για να προωθήσουμε τα εναλλακτικά καύσιμα. Υπάρχει και ένα πακέτο χρηματοδότησης μεταφορών στο μέλλον, αλλά αυτό είναι ένα ξεχωριστό ζήτημα. Αυτή τη στιγμή, ως προς το πακέτο οχημάτων, Ε, θα υπάρξουν μέτρα ως προς τις δημόσιες μεταφορές και τις δημόσιες μετακινήσεις προσπαθούμε να λάβουν υπόψη τις βέλτιστες ε, τακτικές. Προσπαθούμε να έχουμε έναν πράσινο τομέα δημόσιων προμηθειών. Είναι στο μέσο ο οποίος ε, είναι καρποφόρος, ιδιαίτερα για τις δημόσιες μεταφορές, σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης. Αυτή την οδό θα ακολουθήσουμε, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε και την οδηγία για τα καθαρά οχήματα. Αυτά είναι τα δύο μέτρα. Θα θέσουμε σε εφαρμογή αυτή την οδηγία. Τώρα, κατά πόσο ήρθα σε επαφή με υπουργούς και πρωτεύουσες. Θα μιλήσω πάλι αγγλικά προς τον κύριο Σάλτε Μόζε, ο οποίος είναι απόν. Συζητώ μαζί τους σε καθημερινή βάση. Υπήρχε μία επιχείρηση που ήρθε σε επαφή μαζί μου. Δεν θα ήθελα να σας μιλήσω για το ποια βιομηχανία αυτοκινήτων ήταν, αλλά με βάση την πρότασή μας για τα βαρέα οχήματα είχαμε μία πολύ σκόπιμη συζήτηση για τα βαρέα οχήματα από συγκεκριμένες βιομηχανίες οι οποίες εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία συζήτησης ενεργά. Ως προς τις απαγορεύσεις διζελοκίνητων οχημάτων στις πόλεις δεν έχουμε σχέδια για μια εναρμονισμένη ευρωβινιέτα. Δεν μας είχε απασχολήσει μέχρι τώρα. Και όπως θα γνωρίζετε, ίσως, αν και κατανοώ το σκεπτικό της απαγόρευσης διζελοκίνητων οχημάτων στις πόλεις, λυπάμαι γιατί αυτοί που καταβάλουν το τίμημα είναι οι κάτοχοι αυτοκινήτων. Αυτοί καταβάλουν το αντίτιμο και όχι οι βιομηχανίες, αλλά οι κάτοχοι οχημάτων. Όπως είπα πολλές φορές, αυτοί που αγόρασαν τα αυτοκίνητα με αυτό το λογισμικό αναστολής βασίστηκαν στην αυτοκινητοβιομηχανία. Άρα δεν φταίνε οι ίδιοι. Γιατί θα πρέπει να υφίστανται τις κυρώσεις με τα νέα κριτήρια εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, με αυτό το νέο πακέτο του Νοεμβρίου, στέλνουμε το σωστό μήνυμα ως προς τα οχήματα, αλλά ως προς τις απαγορεύσεις θεωρώ ότι οι βιομηχανίες καθώς και τα οχήματα που κυκλοφορούν θα πρέπει να μετασκευαστούν πρώτα και μετά να υπάρξει απαγόρευση κυκλοφορίας διζελοκίνητων οχημάτων. Ως, το, ως προς το τέταρτο πακέτο, το οποίο θα εγκριθεί και γιατί έχει καθυστερήσει, Υπάρχουν επιπρόσθετα στοιχεία τα οποία έχουν εισαχθεί στο αρχικό πακέτο και γι' αυτό έχει καθυστερήσει από το Δεκέμβριο μέχρι μάλλον τον Απρίλιο που θα υποβληθεί. Υπήρξαν τεχνικοί λόγοι καθυστερήσεων και όπως σας είπα και πριν θα έχουμε δύο γύρους δοκιμών και επιβεβαιώσεων και ο δεύτερος γύρος εξαρτάται από τις ε, τεχνικές εξελίξεις και έχουμε βεβαίως και τους παράγοντες συμμόρφωσης. Ως προς τη μετασκευή του εξοπλισμού, hardware, Αυτό είναι ένα από τα πλέον σημαντικά ζητήματα, γιατί αυτά τα οχήματα δεν βρίσκονται μόνο στην Ανατολική Ευρώπη. Τα βρίσκεται και σε... Some, ε, areas in Europe. Δεν θα τα βρίσκεται μόνο στις πρώην ανατολικές χώρες, αλλά θα τα βρίσκεται και σε διάφορες ε, επαρχιακές πόλεις της Ισπανίας η Volkswagen παραδέχτηκε ότι θα κάνει αυτή τη μετασκευή hardware, αλλά είναι ιδιαίτερα δαπανηρή. Όχι, όχι για τους καταναλωτές, ελπίζω. Δηλαδή, να μην μετακυλήσουν αυτές τις δαπάνες στους καταναλωτές, κάτι το οποίο θα ήταν ιδιαίτερα άδικο. Γιατί ξέρετε ότι ήταν μια κερδοφόρα εταιρεία, τουλάχιστον μέχρι πέρσι. Δεν θα σας μιλήσω για τις προσωπικές μου απόψεις. Όπως είπα στην εισαγωγή μου, θα προσπαθήσουμε να λάβουμε υπόψη αυτές τις ε, δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, αλλά θέλουμε τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν μαζί μας και θα θέλαμε επίσης τα κράτη-μέλη τα οποία δεν θα πληγούν ιδιαίτερα από το DRC, δεν θα ε, παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλές εκπομπές. Δεν βλέπω ανταπόκριση από τα κράτη-μέλη. Αν και τα κράτη-μέλη αυτά πλήττονται και από το σκάνδαλο Diesel, αλλά και από τους κατασκευαστές. Και φυσικά πλήττονται και από τους ρήπους του περιβάλλοντος. Θα δούμε τι θα κάνει και ο Επίτροπος Βέλα επί του θέματος. Θα το κάνουμε από τη δική μας πλευρά, αλλά θέλουμε και τη συνεργασία των κρατών μελών, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. χρειάζεται πίεση. Όχι σε μας, ξέρω τι εννοείται και στα περισσότερα ζητήματα είμαι με σας, στη δική σας πλευρά. Αλλά τα κράτη-μέλη έχουν μια μεγάλη βιομηχανία αυτοκινήτων, πολλά κράτη, όχι όλα, αλλά θα πρέπει να προβλέψουμε, όχι να αντιδρούμε, γιατί Διαφορετικά σε μερικά χρόνια θα υπάρχει μεγάλη εισρωή οχημάτων, ιδιαίτερα ηλεκτρικών οχημάτων από την Κίνα. Γι' αυτό πρέπει να προβλέψουμε και όχι να αντιδρούμε. Η συνεργασία δεν είναι ικανοποιητική, αλλά το επαναλαμβάνω αυτό εδώ και δύο χρόνια. Δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα τα τελευταία δύο χρόνια. Τώρα το θέμα της Κίνας θα το απαντήσω γραπτός, γιατί δεν είμαι ικανή αυτή τη στιγμή να απαντήσω σε ένα τόσο τεχνικό ερώτημα, προς το παρόν τουλάχιστον. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζουμε ότι όσο θα τους μιλάτε, τόσο περισσότερο θα ανοίγουν τα αυτιά, τα αυτιά τους και θα έχουμε κάποια αποτελέσματα και κάποια δραστηριότητα. Ευχαριστούμε πολύ την Επίτροπο. Κατανοώ ότι τα μέλη μας εκτιμούν ιδιαίτερα αυτή τη συνεισφορά σας. Ευχαριστούμε.